θα νικήσουμε αυτή την κρίση την οποία πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Βαν Ρομπέη. Κλείνει η συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι από αυτού του θέματος. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι δηλώσεις ε, της ε, Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την ε, συνδιάσκεψη κορυφής ε, G20. Και βλέπω τον κύριο Σάστελ, ο οποίος ετοιμάζεται να λάβει το λόγο. And when he takes his seat, I give him the floor straight on. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη συζήτησαν για τους G20 στις 20 Οκτωβρίου και τότε επίκειτο η σύνοδος των G20. Στη συνέχεια είδαμε τι συνέβη στη Σεούλ. Άρα προετοιμαστήκαμε και σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Κατανοήσαμε ότι η έλλειψη συνοχής θα μας οδηγούσε σε έλλειψη αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Και τα σχόλια ολόκληρου του κόσμου ήταν μετριοπαθή σε σχέση με τα αποτελέσματα της Συνόδου της Σεούλ. Θα πρέπει παρόλα αυτά να παραμείνουμε αισιόδοξοι, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν εντυπωσιακά όσο θα επιθυμούσαμε. Ήμασταν πεπισμένοι πριν από την Σεούλ ότι αυτή ήταν μια μεγάλη δοκιμασία. Δεν έπρεπε να χάσουμε την αρχική μας όθηση δεν θα έπρεπε να σφάλουμε σε διεθνές επίπεδο θεωρώντας ότι δεν αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζαμε πριν από ένα χρόνο ή και έξι μήνες. Βεβαίως, οι πολιτικοί αρχηγοί λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της πολιτικής. Όμως φέρουν και μία άλλη ευθύνη, εξίσου σημαντική. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτές οι προσπάθειες να μην παραμείνουν επί χάρτου. Η σύνοδος της Σεούλ κατέδειξε ότι η πραγματική πρόκληση για τους G20 είναι να κατανοήσουμε πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη θέση σε εφαρμογή αυτών των μέτρων. Πώς μπορούμε να περάσουμε σε απτά αποτελέσματα. Και αυτό για δύο λόγους οι αγορές δεν αρκούνται σε δηλώσεις. Έχει σημασία τι θα συμβεί 2, 10 ή 30 μέρες μετά από τη λήξη της Συνόδου, όταν θα διαπιστώσουμε την πραγματική υγεία της οικονομίας, την κατάσταση υγείας της οικονομίας, διότι δεν αρκούμεθα στη, σε μια διήμερη σύνοδο. Τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια και όπως γνωρίζετε αυτό είναι κάτι και το μόνο που θα μπορούσε να ήταν χειροπιαστό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να ασκήσουν έλεγχο και να δώσουν μια πολιτική όθηση στην πολιτική ατζέντα μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων μεταξύ δύο συνόδων και η G20 θα πρέπει να αποτελέσει μία εξελικτική διαδικασία και όχι στιγμιαίες συναντήσεις. Επί της ουσίας βλέπουμε μία αναπτυξιακή πορεία η οποία είναι εξισορροπημένη και βασίζεται σε, ορισμένες, σε ορισμένα συγκεκριμένα πλαίσια, ενός ε, δηλαδή κοινού φορολογικού πλαισίου, ενιαίου φορολογικού πλαισίου και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 ένα πρόγραμμα αναθεώρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται στο peer review μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας της Συνόδου των G20. Ο καθένας θα πρέπει να διαδραματίσει το δικό του ρόλο έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στην αναπτυξιακή αυτή πορεία. Για άλλη μία φορά και μέσα στα πλαίσια των προηγουμένων σχολείων μου πιστεύω ότι η μάχη κατά του προστατευτισμού δεν ε, ε, δεν επιτυγχάνεται μιας διαπαντός. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία επαγρύπνησης. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για την αναθεώρηση μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς ε, Νομισματικού Ταμείου έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει καλύτερα την ε, διεθνή πραγματικότητα και να μπορέσει να βοηθήσει και τις αναδυόμενες ε, οικονομίες. Εμείς μειώσαμε την παρουσία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κρατήσαμε αυτά που επιθυμούσαμε περισσότερο. Δηλαδή να μπορούμε να ασκούμε επιρροή στο διεθνές προσκήνιο. Ε, στη συνέχεια είχαμε τη συμφωνία της Βασιλείας Τρία. δηλαδή τις κεφαλαιοχικές απαιτήσεις των τραπεζών. Κινηθήκαμε προς την σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε πολύ σωστά τη Συμφωνία της Βασιλείας 3. Το θέμα αυτό παραμένει στην πολιτική μας ατζέντα και στην πολιτική ατζέντα των G20. Αν δούμε τι συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τον πόλεμο των νομισμάτων, όπως ε, ονομάζεται, νομίζω ότι ασκήσαμε τη σωστή επιρροή, καταφέραμε πολλά και δεν θα πρέπει να προβούμε σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις νομισμάτων. Η ε, Γαλλία φέρει την ευθύνη της ε, ε, οργάνωσης της επόμενης συνόδου των G20 μετά τη Σεούλ. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε από κοινού με συντονισμό έτσι ώστε εν τη Συνόδου των Κανών του 2011 να παραμείνουμε στο προσκήνιο και να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς προκλήσεις έτσι ώστε να συνεισφέρουμε και να δώσουμε τη σωστή όθηση για να φτάσουμε στους μεσοπρόθεσμους στόχους για να οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή πορεία μέσα στα πλαίσια των διεθνών αγορών και να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε καλύτερα το σημερινό κόσμο μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι G20 θα πρέπει να καταδείξουν το επόμενα χρόνια ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά πρωτίστως πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος κ. Μπαρός, εκ μέρους της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η συνάντηση κορυφής που έλαβε χώρα αυτό το μήνα ασχολήθηκε με το εξής. Εφόσον υποχωρεί η κρίση, η G20 θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο συντονισμό. Μετά την συνάντηση κορυφής αυτού του μήνα, μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι υπήρχαν τα διάφορα αρνητικά σενάρια παλαιότερα, τα οποία όμω δεν επιβεβαιώθηκαν. Βλέπουμε ότι η G20 περνάει σε μια πιο σταθερή ε, στάση και παρά τις συζητήσεις και παρά το γεγονός ε, ότι η φορολόγηση παραδείγματος χάνει ένα θέμα επί το οποίο δεν υπήρξε συμφωνία η G20 και πάλι εξέπεμψε ένα σημαντικό μήνυμα αποφασιστικότητας ε, σταθερή πρόοδος για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις ξέρω ότι τα αποτελέσματα αντιμετωπίστηκαν με κάποια επιφυλακτικότητα γιατί δεν ήταν θεαματικά δεν υπήρξε την τελευταία στιγμή κάποια ουσιαστική πρόοδος αλλά αυτό που δεν μοιάζει να γίνει κατανοητό ακόμα και από τους σκεπτιστικιστές είναι ότι και μόνο αυτή η συνάντηση G20 είναι ένα θεματικό γεγονός. Δεν πρόκειται απλά για άλλη μια διαδικασία όπου όλοι ε, εκφράζουν τις απόψεις τους και καταλήγουν σε συμβασμούς. Εκτός λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έστειλε τα δικά της τα μέλη, οι χώρες του G20 ε, ε, συμπεριλαμβάνουν τι ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Αργεντινή, την Νότια Κορέα, την Νότια Αφρική και το γεγονό και μόνο ότι όλοι αυτοί εμπλέκονται σε μια διαδικασία για να αντιμετωπίσουν τι παγκόσμιε ανισορροπίε και συμφωνούν, παραδείγματο χάρη, για χρηματοπιστωτικού κανονισμού και μόνο το γεγονό αυτό πρέπει να τύχει αναγνώριση. Τεράστια λοιπόν πρόοδο, η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από κάποια χρόνια η συνάντηση ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία και ε, υπήρξε πλέον μια νέα ε, ημερήσια διάταξη. Δεν ήταν ένα γεγονό ε, που απλά ήταν σημαντικό. Εστέφτη λοιπόν επιτυχία και οι Ένωση που εκπροσωπήσαμε εγώ και ο πρόεδρο, ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εμεί συνεισφέραμε σημαντικά και σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Επίτροπο κύριο Όλι Ρεν, που είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Σε γενικέ λοιπόν γραμμέ, τα συμπεράσματα αντικατοπτρίζουν τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη Σεούλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να είναι ε, πολύ περήφανη για την σημαντική τη συνεισφορά στη διαδικασία αυτή. Και θα σα ε, παραθέσω κάποια σημαντικά επιτεύγματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούσε η συνδιάσκεψη να σημειώσει πρόοδο στο πώ είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιε ανισορροπίε και οι εντάσει που υπάρχουν. Γνωρίζαμε όλοι μας ότι θα ήταν ένα Ηράκλειο έργο το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανισορροπίες. Όμως η G20 μετά από σκληρές ε, και ε, κοπιώδεις διαβουλεύσεις δρομολόγησαν ένα μηχανισμό ο οποίος θα συνενώνει όλους τους μηχανισμούς για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Όσοι μετέχουν στην G20 κατόρθωσαν να περιορίσουν τις ανισορροπίες και να διατηρήσουν τις ανισορροπίες σε επίπεδο ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Οι της G20 και το πώς να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες κατέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, περάσει στην άλλη πλευρά, έχει περάσει τα τεράστια προβλήματα. Ε, οι ηγέτες των G20 πράγματι ίσως είναι καλύτεροι για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες ανισορροπίες. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία για να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες και αυτά βρίσκονται στη βάση του μηχανισμού των G20, ο οποίο θα αρχίσει να ισχύει στα μέσα του 2011. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει πριν από την επόμενη συνάντηση που θα λάβει η χώρα τον Νοέμβριο του 2011. Τώρα λοιπόν εστιάζουμε την προσοχή μα στην ενίσχυση αυτού του μηχανισμού στο βαθμό του δυνατού για να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζεται σωστά κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Προεδρία στου G20 το 2011. Τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά συμφωνώ βέβαια ότι τώρα πλέον οφείλουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Το δεύτερο επίτευγμα έχει σχέση με ε, τις ε, ε, συναλλαγματικές ισορροπίες. Και πάλι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στο να υπάρξουν κάποιες λύσεις συνενετικές. Προχωράμε περισσότερο ε, προς ένα σύστημα ισοτιμιών, συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα είναι προσαρμοσμένο στην αγορά. Συμφωνήσαμε επίσης ότι δεν πρέπει να προβαίνουμε απαραίτητα σε υποτιμήσεις και να υπάρχουν κάποιες ανισόρροπες τάσεις στις ισοτιμίες. Η Γαλλική Προεδρία θα ασχοληθεί με μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Επίσης, με χαρά μου, η G20 είδα ότι επικύρωσαν την ιστορική μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είχαμε ξεπεράσει, ξεπεράσαμε μάλιστα και τις προσδοκίες και αυτό το κατορθώσαμε χάρη σε μια ανοιχτή προσέγγιση των μελών των G20. Όλοι έχουμε την ευθύνη ε, για τα τεκτενόμενα, άρα δηλαδή και το Διεθνές Ταμείο πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ε, τα καθήκοντα που του έχουν τεθεί, που αφορούν κυρίω τις ανισορροπίες. Οι αναδυόμενε οικονομίε πρέπει να αποδείξουν ότι και αυτέ ε, θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο, βέβαια, αλλά θα αναλαμβάνουν και μεγαλύτερες ευθύνε όσον αφορά την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Ένα τέταρτο επίτευγμα τη διακυβέρνηση ήταν να διατηρηθεί ο ενθουσιασμό για μεταρρυθμίσει και να εφαρμόζονται τα αποτελέσματα. Η Βασιλεία 3 μεταρρύθμιση, το χαιρετίζουμε και η G20 θα συνεχίσει ε, να αναζητά τους απαραίτητους θεσμούς. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες σε πλαίσιο μακροοικονομικό, ε, στο shadow banking, ε, στην αγορά των παραγόγων και στην αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται σε πάρα πολλά αυτά τα θέματα και οι εσωτερικές διεργασίες θα ενταχθούν στην διαδικασία των G20. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την σωστή ε, συνεπή εφαρμογή όλων αυτών των δεσμεύσεων σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο επί του οποίου έχουμε συμφωνήσει και να διασφαλίζουμε και ίσους όρου ανταγωνισμού. Οι ΗΠΑ Πολιτείε μα διαβεβαίωσαν ότι συμμερίζονται τη δική μα την αποφασιστικότητα. Επίση, στη Σεούλ μπορέσαμε ε, να επιτύχουμε και νέο ενθουσιασμό, δέσμευση των G20 να ε, καταπολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον προστατευτισμό. Επίσης, με την συνένεση που προέκυψε από τη Σεούλ όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη κατορθώσαμε να την εντάξουμε στη μερίσια διάταξη των G20. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των δωρητών και το σύστημα των Ηνωμένων ε, εθνών. Θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους της χιλίτιας και όλα αυτά συμβαδίζουν με τις ε, προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική αυτή. Η πράσινη βίβλος της Επιτροπής έχει τεθεί πλέον προς διαβούλευση και περιμένω τη δική σας την συνεισφορά. Και τέλος χαιρετίζω την δέσμευση των G20 για τη διαφθορά για παρεμφερή θέματα στο μέλλον δεν θα πιστεί κανείς ε, κόπου και χρόνου για να συμμετέχει αποτελεσματικότερα στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο Κανκούν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, η ανάπτυξη που δείχνουν οι επιχειρήσεις δείχνει ότι το G20 έχει πλέον καθιερωθεί ως το μεγάλο φόρουμ της ε, οικονομίας. Συμμετείχα και στο G20 Business Summit το επιχειρηματικό φόρουμ όπου ασχολήθηκε και με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Επίσης η Ευρώπη, η Βόρεια και Νότια Αμερική και η Ασία ε, συναντήθηκαν με μια αντιπροσωπεία στην οποία ε, στην οποία συγγύθηκε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και έγινε πρόταση η Ευρώπη να ε, έκανε πρόταση η Ευρώπη να ενταχθεί η κοινωνική διάσταση και οι συνθήκες εργασίας στο, στα στο σχέδιο ε, των ε, ε, συμπερασμάτων. στην επόμενη φορά θα έχουμε ένα από τα κράτη-μέλη στον φάλαμο καθοδήγησης η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να στηρίξει πλήρως την Γαλλική Προεδρία και τις προτεραιότητές της. Μία από τις οποίες είναι η μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος έτσι ώστε να βελτιωθεί η σταθερότητα και να, μειωθούν οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών και βεβαίως αυτό αφορά και τις διακυμάνσεις των τιμών πρώτων υλών. Η Κομισιόν θα ενισχύσει ε, την αγορά πρώτων υλών πάσης φύσεως ε, το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά ε, το γεγονός ότι η Γαλλική Προεδρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Κομισιόν, για την Ευρώπη να αφήσει το αποτύπωμά της στο μέλλον. Η Ευρώπη θα ενισχύσει τη θέση της στο επίκεντρο του οικονομικού του Παγκοσμίου Οικονομικού Συστήματος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci. Thank you, President ε, ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο κύριο Μπαρόζο. Τώρα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και πρώτα απ' όλα ο κύριος Γκοζέ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι διαθέτω ένα λεπτό. Κύριε Προεδρεύοντα, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα καταρχήν, κύριε Προεδρέποντα, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι εκτίμησα την ε, διαυγή παρουσίασή σας των αποτελεσμάτων της Συνόδου των G20 και συμμερίζομαι και την στάση σας για το μέλλον. Τα αποτελέσματα ήταν σχετικά αδύναμα παρόλο που εγκρίναμε την ε, Συμφωνία της Βασιλείας 3 και παρά την αναθεώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βλέπουμε ότι οι προτάσεις της σεούλ είναι φιλόδοξες αλλά και επίγουσα σημασίας για να αντιμετωπίσουμε τη δυσχερή παρούσα κατάσταση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει σωστά το ρόλο της γιατί διαθέτει ειδικό βάρος. Είπατε ότι οι συμπολίτες μας περιμένουν δράση και όχι δηλώσεις επί χάρτου. Η κατάσταση της οικονομίας οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης διεθνών κανόνων. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι αφελής, θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαιότης. Ο κύριος Μπούλμαν, ο οποίος έχει δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Χάρμς ε, σήμερα το πρωί ε, στη συζήτηση που έγινε έθεσε το ερώτημα γιατί πλέον ε, οι σύνοδοι αυτές δεν εμπνέουν τους πολίτες γιατί από αυτές δεν απορρέει η αισιοδοξία. Ακούγοντας λοιπόν εσάς σήμερα το πρωί αλλά και τώρα κύριε Μπαρόζο, κύριε Βάνο Χομπέι και ακούγοντας και το Συμβούλιο καταλαβαίνω πρέπει να σας πω γιατί δεν μεταδίδεται αυτός ο ενθουσιασμός και ούτε καν και στην αίθουσα δεν υπάρχει ενθουσιασμό, Για δέστε λιγάκι εδώ τα άδεια έδρανα. Θα ήταν πολύ πιο σημαντικό αν ήταν εδώ παρόντε συνάδελφοι. Γιατί δεν είναι παρόντε, λάθο βέβαια που δεν είναι εδώ. Όμω, ε, ακόμα και αν ήταν εδώ δεν θα ενημερώνονταν για κάτι το καινούριο. Μα λέτε πράγματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει 20 φορέ εφημερίδε και δεν δίδεται καμία απάντηση σε αυτό το οξύ ερώτημα που ετέθη. Τι θα γίνει τελικά με το φόρο συναλλαγματικών, ε, φόρο ανταλλαγών, συναλλαγματικών ανταλλαγών το θέμα αυτό ε, δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου των και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί. Να γνωρίζω επίσης γιατί η Βελγική Προεδρία λέει ότι ε, τάσεται υπέρ αυτού του φόρου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις τελευταίες τρεις συναντήσεις του απλά είπε ότι θα πρέπει να γίνει μία μελέτη σκοπιμότητα σε παγκόσμιο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνετε στο Συμβούλιο ότι στο θέμα αυτό οδηγείστε σε αδιέξοδο και κύριε Μπαρόζο στις αρχές αυτού του έτους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνει μελέτη σκοπιμότητας ξεχωριστά για την Ευρώπη. Εάν λοιπόν πείτε μια άποψη επ' αυτού θα γεμίσει η αίθουσα και θα σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Όμως πλέον μην υπεκφεύγετε γιατί μόνο για την Ευρώπη μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ρωτήστε λοιπόν τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προπλογισμών με τι είδους αμεληταία ποσά είναι αναγκασμένοι να τσακώνονται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν τους ρόλους να του ενσαρκώνει κανεί σωστά και εφόσον γίνεται αυτό, τότε πράγματι θα γεμίσουν οι αίθουσε, θα υπάρξει ενθουσιασμό και εμεί αυτό περιμένουμε από εσά. Κυρία Ντεσάντ, εκ μέρου των Φιλελευθέρων, δύο λεπτά. Εάν η Ευρώπη δεν έχει μία κοινή πολιτική, ένα κοινό ε, όραμα, τότε η επόμενη ε, G20 θα είναι μία ανταλλαγή πυρών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις δικές της δυσκολίες και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα διανύει μία δυσχερή περίοδο και έτσι υπάρχει ένας ανταγωνισμός που είναι αποσταθεροποιητικός για τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι στο G20 θα πρέπει να μιλήσουν για μία νέα διεθνή νομισματική τάξη που να βασίζεται σε ένα καλάθι νομισμάτων όπου θα συμμετέχει και το One και το δολάριο και το ευρώ. Επίσης θα πρέπει να ε, δούμε πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και δεν έχουμε αξιολογήσει τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Μιλάμε για ρύθμιση των αγορών πρώτων υλών σε σχέση με τα ορυκτά και αγροτικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού πρώτων υλών, διότι υπάρχει μεγάλη ένδυα ορισμένων προϊόντων. Εδώ λαμβάνω υπόψη την Κίνα καθώς και την κερδοσκοπία κατά των ε, αγροτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον λοιμό που μαστίζει ορισμένες ε, υποανάπτυξη χώρες. Είμαι πεπισμένη ότι η Γαλλική Προεδρία δεν θα είναι χρήσιμη παρά μόνο εάν εγγράψει αυτή την προσπάθεια σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο κύριος Λεχαϊρίκ, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το εύρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ε, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον απαιτούν αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επίπεδο των G20 που αφορά την, τους κανονισμούς ε, της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς. Δεν θα πρέπει να γίνει ο κόσμος ε, μια καπιταλιστική ζούγκλα, αλλά θα πρέπει να επιβάλλονται πρότυπα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και να υπάρξει απασχόληση. Υπάρχει η μάστιγα της ανεργίας που πλήττει 250 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο λόγω και της ε, ισχύουσας πολιτικής λιτότητας. Θα πρέπει να σταματήσουν οι φορολογικοί παράδεισοι και να υπάρξει ένα σύστημα φορολόγησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και βεβαίως θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε και με τις τιμές πρώτων υλών ξεκινώντας από τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και ένας άλλος ρόλος που θα πρέπει να παίξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα αφορά την, ανάπτυξη ε, την δημιουργία απασχόλησης και βεβαίως θα πρέπει να σταματήσει αυτό το σκάνδαλο των ε, οίκων αξιολόγησης οι οποίοι βεβαίως ε, είναι και κριτές και ελεγχόμενοι. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κυριος Παπανικολάου έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε οι δηλώσει των αποτελεσμάτων της συνόδου g 20 ήταν σίγουρα σημαντικές ωστόσο μια δεύτερη ανάγνωση εγείρει σημαντικά ερωτήματα για συγκεκριμένα σημεία. συγκεκριμένα είκοσι ανεπτυγμένες χώρες απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση σε όσε χώρες εφαρμόζουν μη συντονισμένες οικονομικές πολιτικέ και όλα αυτά την ίδια στιγμή που άλλη οικονομική πολιτική εφαρμόζουν οι ηπα ενισχύοντα τη ρευστότητα άλλοι τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης που επιλέγουν αυτή την περίοδο τη λιτότητα άλλοι η κίνα που επιλέγει να διατηρεί υποτιμημένο το νόμισμά της. επομένως προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα έχει μια τέτοια δήλωση και σε ποιον τελικά απευθύνεται γιατί μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω πως το μήνυμα αυτό έχει αποδέκτη χώρες που έχουν ελάχιστη σημασία στην παγκόσμια οικονομία. αν όμως πάλι η G20 έκαναν μια τέτοια δήλωση με αποδέκτη τον εαυτό του, τότε πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικής συνεννόησης σε μια οικονομική περίοδο που οι αντιδράσεις πρέπει να είναι άμεσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο κύριος Γκόρεντς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Αρχικά θα απίθανε το ερώτημά μου στον κύριο Μπαρόζο, επειδή όμω αποχώρησε το, το απευθύνω στη Βελγική Προεδρία. Σήμερα μπορεί να κάνει κανεί εμπορικό ντάμπινγκ χωρί να παραβαίνει του κανόνε αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ. Με ένα ε, ε, υποτιμημένο νόμισμα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Παρότι σιγά σιγά ασχολούμαστε με το θέμα τη υποτίμηση και της ανταγωνιστικότητας. Το θέμα που είναι, απαράδεκτο, που είναι βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να τίθεται. Λοιπόν, στρέφουν προς βελγική κυβέρνηση και λέω, αν οι G20 δεν μπορούν να βάλουν μια τάξη στην νομισματική αταξία, πιστεύετε ότι ο ΠΟΕ θα μπορέσει να βγει άφικτος από αυτή τη διαδικασία. Merci. Mr. Ε, ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σύνοδος των G20 του Νοεμβρίου κατά την άποψή μου δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα κύριε πρόεδρε. απέδειξε για άλλη μια φορά τη δεσπόζουσα θέση των ηνωμένων πολιτειών και την προσπάθεια της κίνας για ουσιαστική αναβάθμιση στο διεθνές στερέωμα. ω γνωστόν η σοβούσα παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 και μετά εκδηλώθηκε όταν οι επενδυτικές τράπεζες στις ηνωμένες πολιτείες η μία μετά την άλλη παρουσίαζαν θέματα ρευστότητος. ως φαίνεται και είναι παγκίνως γνωστόν αναγκάστηκε η κυβέρνηση της αμερικής να εκδώσει νέο χρήμα. το εμφανές είναι στην πρώτη φάση 700 δισεκατομμύρια δολάρια και στη δεύτερη φάση εντελώς πρόσφατα άλλα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. σε αντίθεση με την συμπεριφορά αυτή στο νομισματικό θέμα των ηπα η ευρώπη και ιδιαίτερα η ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στην αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην αυστερώς ελεγχόμενη νομισματική πολιτική με αποτέλεσμα να αφήνει χώρο στις αγορές για κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των λιγότερων ανθεκτικών ε, οικονομιών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης. Προτείνω κύριε Πρόεδρε να μελετηθεί το θέμα εκδόσεως νέου χρήματος, νέου χρήματος στην Ευρώπη είτε με τη μορφή ε, ε, bank notes είτε με τη μορφή ευρωομολόγου. Ευχαριστώ πολύ. please. Mr. Ευχαριστώ. Μας περιμένουν οι συμπολίτες, περιμένουν από την Ευρώπη ε, να αποφανθεί για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα πρέπει να είμαστε μία δύναμη λήψης απόφασης, αποφάσεων. Πολλοί τόνισαν ότι η Γαλλική Προεδρία του G20 θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για την Ευρώπη. Συμμερίζομαι αυτή την άποψη και νομίζω ότι θα ήταν ε, σκόπιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πληροφορείται για τις εξελίξεις συζητήσεων στους G20. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα εκφραστεί ενώπιον μας και ελπίζω να, γίνει αυτή η... να εισακουστεί αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Και τώρα για να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές, δίνω το λόγο καταρχήν στον, πρόεδρο, στον Επίτροπο Πίμπαλξ. Πρόεδρε, η ε, G20 είναι μια ειδική σύνοδος ε, και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Η διαδικασία βέβαια ε, είναι ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από αυτά τα θέματα που συζητήθηκαν. Πρόκειται για την φορολόγηση του χρηματοψηφιστικού τομέα. Ακόμα και αν δεν υπήρξε κάποια τομή, ε, συμφωνήθηκε να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα αυτό υπό τη Γαλλική Προεδρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να στηρίξει την εργασία των G20 που αφορά ε, στην εξέταση του φόρου διατραπεζικών συναλλαγών. Όπως σας είπα, η G20 δουλεύει με τη συνένεση και πάρα πολλά μέλη των G20 σε αυτή τη φάση δεν συμμερίζονται τις απόψεις μας επί του θέματος. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη συνένεση. Εν τω μεταξύ πρέπει να αναζητήσουμε και άλλες διασφαλίσεις ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέα συνεισφέρει δίκαια μέσα από ε, μέτρα όπως είναι πραγματικό φόρος επί των ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων και συναλλαγών. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδρομή και τους στόχους, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε γρήγοροι, σίγουροι ότι ο χρηματοψηφιακός τομέας συμβάλλει σημαντικά στα δημόσια οικονομικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, κυρίως για την στήριξη που του προσφέρθηκε κατά διάρκεια της κρίσης. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μορφή φόρου επιβάλλουμε θα αποφέρει και ωφέλει, θα αυξήσει τα έσοδα χωρίς να ε, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτό το μοσαϊκό των διαφόρων φόρων που υπάρχουν επί του εξωτερικού τομέα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αποτελούν εμπόδιο για την κοινή αγορά. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει δύο προσεγγίσεις για το φόρο αυτό. Πρώτον, ε, φόρος ε, ε, χρηματοψητικών δραστηριοτήτων. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να χρηματοδοτούνται τα κέρδη γιατί με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο θα αποφέρει και εισόδημα. Και επιπλέον ο φόρος αυτός ε, δεν θα είναι τόσο ευάλωτος και εκτεθειμένος απέναντι στους κινδύνους της ανταγωνιστικότητας, πράγμα που ισχύει για άλλα είδη φόρων. Ένας τέτοιος λοιπόν φόρος συναλλαγών θα πρέπει να προαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε τους στόχους μας σε τομείς όπως είναι η αναπτυξιακή βοήθεια και η αλλαγή του κλίματος. Με την σωστή επιλογή του είδους του φόρου και την εφαρμογή του θα μπορούσαμε να έχουμε μια σημαντική πηγή εσόδων και να διατηρήσουμε παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει, επιθυμεί να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο και να καταθέσει πρωτοβουλίες το 2011. Το πρώτο βήμα θα είναι μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων για την περίπτωση εφαρμογής του φόρου, κάτι που θα καλύπτει όλα αυτά που είπαμε. Και εκεί θα λάβουμε επίσης υπόψη μας και τις αναλύσεις των κρατών μελών. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στον, ε, στους ε, φορείς ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αυτό είναι σημαντικό πριν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση. Και εγώ από δική μου πλευρά, κύριε Πρόεδρε, θέλω επίση να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η σύνοδο των G20 ε, στην ημερήσια διάταξη συμπεριέλαβε ε, στόχου ανάπτυξη ε, με αποφασιστικότητα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν τελικά να αποβούν προ όφελο των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πίτροπο και ο κύριος Σάστελ θα λάβει το λόγο εκ μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένα κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι γενικά ε, πριν από τη σύγκληση της Συνόδου των G20 θεωρούσαμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση φτάσαμε σε αποδεκτά αποτελέσματα σε αρκετά ζητήματα και θα θέλαμε οι G20 να παραμείνουν ένα αξιόπιστο και θεμητό φόρουμ που να μπορέσει να δώσει μία όθηση σε όλα μας τα ζητήματα εν ώψη της παγκοσμιοποίησης έτσι ώστε να εισακουστεί η φωνή των Ευρωπαίων. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες, αναφερθήκατε σε αυτές αλλά θεωρούμε ότι ήταν η ικανοποιητική η διαθεσμική συνεργασία που ε, έφτασε, που οδήγησε στις, στις εργασίες του G20. Πρόκειται για την πέμπτη διάσκεψη μέσα σε δύο-δυόμιση χρόνια. Φτάσαμε σε μία χρηματοοικονομική σταθερότητα, σχετική σταθερότητα, αλλά φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ε, αναγνωρίζω αυτά που μας είπε η Επιτροπή σε σχέση με τον φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τον ε, φόρο αυτό, το διατραπεζικό φόρο συναλλαγών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Ως προς αυτή τη διατραπεζική εισφορά πιστεύουμε ότι ότι ε, δεν υπάρχει συμφωνία ούτε ως προς το στόχο ούτε ως προς την χρήση αυτής της εισφοράς, των εσόδων δηλαδή που απορρέουν από αυτή την εισφορά. Και νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία, εθνικά στοιχεία που διαφέρουν. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος παρονομαστής και να φτάσουμε σε μία εξυγίανση των τραπεζών η οποία θα ε, οδηγήσει στην αντιμετώπιση των κρίσεων με βάση την νομοθετική πρόταση της ε, Επιτροπής. Με αυτά τα δεδομένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου συμφώνησε ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τα καθεστώτα διατραπεζικών εισφορών και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα φτάσει σε συμπεράσματα πριν από την διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου. Ως προς αυτό το διατραπεζικό φόρο, τη διατραπεζική εισφορά, το ΕΚΟΦΗΝ θα εξετάσει πώς μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές εναλλακτικές για να αποφύγουμε τις ε, φοροδιαφυγές και να πατάξουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σάστελ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα τη συζητήσεις, αλλά σας παρακαλώ μην φύγετε από την αίθουσα, διότι τώρα περνάμε στην, στην τελετή απονομής των βραβείων Λουξ. Σας ευχαριστώ.